οι περικοπές σε αυτό το τομέα και ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη απορρόφηση των πιστώσεων. Ο τομέα τον οποίο πρέπει να, προσέξουμε είναι τα απορροκυπευτικά. Ε, έγινε μία συμφωνία στον τριμερή διάλογο ε, για το φετινό προϋπολογισμό 2012 όπου επαναφέραμε τους αριθμούς της Κομισιόν και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Ε, προσθέσαμε μία παρατήρηση ότι η διαφορά αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουμε τις οργανώσεις παραγωγών και τον ε, τομέα. Περιμένουμε ακόμα συγκεκριμένε προτάσεις από την Κομισιόν για το πώς ε, θα χρησιμοποιήσουν αυτό το συγκεκριμένο κονδύλι προς αυτό το συγκεκριμένο σκοπό και θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις και πρέπει επίσης ε, να δούμε εάν πρέπει το 2013 να προσαρμοστεί αυτός ο τομέας αλλά θα ήθελα να ξέρω πρώτα τις απαντήσεις αυτού του έτους, του προπορισμού αυτού του έτους διότι αναμένουμε πληροφορίες από την Κομισιόν. Τέλος, τα πιλωτικά προγράμματα. Είπα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ότι ε, θέλω να προτείνω προγράμματα ανάπτυξης, ε, τα οποία υποστηρίζουν πολλές ομάδες, αλλά κάταρχας, παρακαλώ, παρακαλώ, ε, μπορεί, κάντε ησυχία, προσπαθώ να τα πω σύντομα, αλλά θέλω ησυχία. Λοιπόν, τα πιλωτικά προγράμματα πριν ε, στοχεύσουμε στα καινούρια και επειδή έχουν ακουστεί πολλές επικρίσεις από το σώμα για παρελθόντα πιλωτικά προγράμματα τα οποία δεν υλοποιήθηκαν και ήταν πιλωτικά προγράμματα τα οποία ήταν προγράμματα κλειδιά για την Επιτροπή μας. Ε, παραδείγματος χάρη το θέμα των περιθωρίων δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα. Γι' αυτό θέλουμε να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές για την απλούστευση της πολλαπλής συμμόρφωσης μέσα στα πλαίσια της, της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Δεν έχει υλοποιηθεί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και θέλω να ξέρω τους λόγους και πρέπει να ξέρει η Κομισιόν ότι είναι ακόμα θέμα προτεραιότητας για μας. Όπως και το ε, θέμα της κερδοσκοπίας ε, και της ε, βάλου φύσης ε, των αγροτικών αγορών. Και πέραν αυτού με την έγκρισή σας θα ήθελα να προτείνω πιλωτικά προγράμματα όπου θα ενημερώνουμε τους παραγωγούς καλύτερα πώς θα αντιποκρίνονται σε αυτή την ευάλωτη φύση των αγορών. Μπορείτε να επικρίνετε το ευάλωτο των αγορών αλλά, ε, και τις διακοιμάνσεις, ε, αλλά πρέπει να έχουν καλύτερη ενημέρωση οι παραγωγοί για να μπορούν να αντιδράσουν και όχι ακαδημαϊκά αλλά πρακτικά. Για αν συμφωνούν οι συνάδελφοι αυτό θα είναι ίσως κάτι ενδιαφέρον ως πιλωτικό πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω προς το παρόν ώσπου να ακούσω την Κομισιόν και τους συναδέλφους. Αλλά χάνουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ο Τζορτζ Λάιον. Θα είμαι και εγώ σύντομος. Σύμφωνο με την προσέγγιση της Έστερ για τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την άποψή της ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση και να αντιδράσουμε αντίστοιχα στις προτάσεις της Κομισιόν. Ε, χρειάζομαι ορισμένες διευκρινήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μπορεί η Κομισιόν να μου διευκρινίσει. Πέρσι είχαμε ένα κονδύλι 10 εκατομμύρια το οποίο δεν μπόρεσε να διαθέσει η Κομισιόν για την ανάπτυξη της υπαίθρου δεδομένου ότι δεν έφτανε ο προϋπολογισμός. Δεύτερον, το 4,5% ε, ε, δαπάνες, ε, επιπλέον δαπάνες για την ύπεθρο, την ανάπτυξη της Επέθρου. Πόσο σαφείς είσαστε για το ποσοστό αυτό είναι εκτιμήσεις, βασίζεστε σε εκτιμήσεις. Δεδομένου ότι τώρα ολοκληρώνεται, φτάνει προς το τέλος του το πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου, ε, διότι πολλές ε, φορές ε, το πρόγραμμα αυτό δεν οδηγείται από τις απαιτήσει, από τα αιτήματα όσο τα διαφορετικά ταμεία. Δεν κατευθύνεται. Ευχαριστώ η Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Έστερ για την καλή της εργασία. Γενικά πιστεύω ότι είναι σωστό η Κομισιόν θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει ε, τομείς εξοικονόμησης αλλά πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν συνάδει με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ιδίω σε, περιοχή, σε περίοδο κρίσεων, ε, πρέπει να προωθήσουμε αναπτυξιακές επενδύσεις. Ε, μέσω του δεύτερου πυλώνα, όπου ο οποίος καλύπτει την ανάπτυξη της υπαίθρου, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, αναπτυξιακή κατεύθυνση για, την, για πρόσθετη αξία. Ορισμένα πιλωτικά προγράμματα δεν υλοποιήθηκαν, ε, το είπε και η Έστερ, ε, γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε ώστε τα προγράμματα τα οποία έχουμε προτείνει εμείς ε, να μην κολλήσουν. Αναφέρθηκε η συγγήτρια στα προκυπευτικά και αν γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να υποδείξουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς που έχουν μαζικά προβλήματα όπως τα γαλακτοκομικά όπου η παραγωγή γάλακτος υποφέρουν διότι αυξάνεται συνεχώς το κόστος παραγωγής και ενοικίασης των μονάδων θέλω να δώσω το λόγο κατευθείαν ε, στη Στή και κατόπιν ε, στην Έστερ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντελάνγκο για την εξαιρετική έκθεση, για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που διαβάσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα περιοριστώ λοιπόν και εγώ στο να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτηματικά που τέθηκαν ε, παρά να κάνω μια παρουσίαση συμπληρωματική της ε, πρότασης προϋπολογισμού μας. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση για το πρόγραμμα γάλακτο στα σχολεία. Διανομής γάλακτο στα σχολεία. Η Κομισιόν έκανε μία πρόταση βάση μιας ε, εις βάθος ανάλυσης της ανάγκης του προπολογισμού των δημοσιονομικών αναγκών. Το 2011 η εκτέλεση αυτού του προγράμματος έφτανε στα 64 εκατομμύρια ευρώ. Και εμεί αυτό που προβλέπουμε για το 2012 βάσει διαθέσιμων δεδομένων δεν είναι μία εκτέλεση που θα πήγαινε πολύ πέρα αυτού του ποσού. Αυτά τα 64 εκατομμύρια ε, τα είχαμε ήδη καταγράψει για το 2011 αλλά με κάποια απογοήτευση και πικρία διαπιστώνουμε ότι τα 90 εκατομμύρια που είχαν προβλεφθεί από τον προϋπολογισμό του 2012 δυστυχώς ούτε φέτος ε, θα φτάσουμε σε αυτό το ποσό. Γιατί σε ένα πνεύμα γενικού περιορισμού των προτάσεων περιπολογισμού αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο μία μικρή αύξηση στα δεδομένα του 2011, δηλαδή ε, προτείναμε απλώς 66 εκατομμύρια. Δύσκολο είναι να δώσουμε μία εξήγηση. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη που δεν ήρθαν να μας παρουσιάσουν πιο ουσιαστικά προγράμματα. και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορούν να συντρέχουν συνθήκες για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Και βεβαίως η κυρία Ντελάνγκε θα μπορούσε να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οποροκυπευτικά. Είναι μια μεγάλη ανησυχία του Επιτρόπου με αυτού και ξέρετε ότι οι υπηρεσίες μας ε, παρακολουθούν πολύ προσεκτικά αυτή την ευαίσθητη αγορά. Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όταν ε, δημιουργείται συνθήκες κρίσης σε αυτή την αγορά για να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα μέσα και να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στις ε, καταστάσεις που θα προκύψουν. Όπως σας είπα, πρόκειται για έναν ευαίσθητο τομέα, για ένα δύσκολο τομέα. Και πραγματικά ε, δίνουμε όλοι μας την προσοχή εκεί. Και θέλω να επισημάνω ότι πέρσι καλωσορίσαμε τη δήλωση ότι αυτό το κοινοβούλιο που υιοθέτησε αυτό το κοινοβούλιο και που συνόδευε τις τελικές αποφάσεις του προπολογισμού πέρσι. Ελπίζω ότι θα μπορέσει και στο μέλλον να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση για να υποστηριχθεί ένας τέτοιος τομέας. Και τώρα, φτάνουμε σε ένα ζωτικό θέμα. Um, so Λοιπόν, τα πιλωτικά σχέδια. Υπάρχει μία σειρά στοιχείων που ήθελα να παρουσιάσω στην κυρία Ντελάνκια, αλλά δυστυχώ ε, δεν έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ παρουσία όλων. Αλλά εγώ είμαι στη διάθεσή σα για να παρουσιάσω όλα τα στοιχεία που θέλετε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Διευθυντά, αλλά με το προηγούμενο θέμα ξεπεράσαμε του χρόνου. Έστερ. Yes, very short, uh, because this... πάρα πολύ σύντομη Βλέπετε το πρόβλημα όταν δεν τηρούμε τα ωράρια. Εργάζονται οι γονείς, τι να το κάνουμε το παιδί. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπάθησε να μας εξηγήσει επακριβέστερα το περιεχόμενο του πιλωτικού προγράμματος. Ξέρουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για αυτό το θέμα, ας τα πούνε μεταξύ τους σε μία ε, σύσκεψη για να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά που είπαν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, ναι, όταν αναφέρεται κάποιο σε ένα τομέα πρέπει να αναφέρεται και σε άλλους, αλλά όταν σας μιλάω για τα, τα, γαλακτοκομικά και αυτά που γίνανε πριν από λίγα χρόνια, εννοώ ότι ε, το έχουμε ξαναντιμετωπίσει το θέμα. Δεν πρέπει να χάνουμε την εστίαση αναφερο, ε, αναφερόμενη σε υπερβολικά πολλούς τομείς. Θα λάβω υπόψη παρατηρήσει των συναδέλφων και του Τζολάινε και άλλων. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ Έστερ, Σα ευχαριστώ όλου. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρία σα. θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στι 3.